Aber ich darf Ihnen sagen, ich bin sehr glücklich und äh, darf das auch für José Manuel Fernández erklären, dass wir als Μιλήσω και εκ μέρους του κυρίου Φερνάντε, ο οποίος ήταν και ο συνεισηγητή. και θεωρώ ότι πραγματικά είχαμε ιδιαίτερα αγαστή συνεργασία. Πολύ καλό το πνεύμα συνεργασίας και αυτό που τελικά κατορθώσαμε είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδιώξουμε να έρθουν πολλές επενδύσεις, να εξυγχρονιστεί η διοίκηση, να βελτιωθεί η διοίκηση και με τον τρόπο αυτό οι πολίτες ε, να μπορούν να εργάζονται με καλύτερο τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν για άλλη μια φορά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και επιτρέψτε μας ε, πριν από την ε, ψηφοφορία να κάνουμε και μία διευκρινήση σχετικά με το νομοθετικό κομμάτι. Κάτι το οποίο έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας οι πολιτικές ομάδες. Θα επανέλθω από αυτού. Ο κύριος Φερνάντες, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα στα Πορτογαλικά. Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, Σκιώδη Συγητή για το έργο του. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμβούλους, τα μέλη της γραμματείας. Ξέρω ότι επιτελέσαμε πολύ σημαντικό έργο. Πήραμε ό,τι καλύτερο από τον καθένα. Και έτσι καταλήξαμε σε ένα τελικό αποτέλεσμα το οποίο είναι πραγματικά καλύτερο από το αρχικό κείμενο. Προχωρήσαμε και σε διάφορες συμβαστικές τροπολογίες, οι οποίες προσπαθούν να συγκεράσουν τις διαφορετικές απόψεις. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους συναδέλφους για τις τροπολογίες τους. Ευχαριστώ λοιπόν όλους σας, τίποτα άλλο. Πρόεδρος, εκ μέρους των συνεδέρφων. θέλουμε και εμείς να σας ευχαριστήσουμε και να σας συγχαρούμε για το έργο σας. Οπότε τώρα θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Προηγουμένως όμως να δοκιμάσουμε ε, τα μηχανήματα. Οπότε παρακαλώ δοκιμαστικά βάλτε τις ε, κάρτες σας, το μηχάνημα για να δούμε. Θα κάνουμε σαν να ψηφίζουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Θα μου τη φέρουν την κάρτα μου. Δεν την έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή, Πρόεδρε. Λέω ο κύριος Ντεπρέ. Πέρα στις ψηφοφορίες λείπουν τρεις ψήφοι. Σύμφωνα με τη δοκιμή αυτή. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν την έκθεση εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Συμβαστική τροπολογία Α, α, υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Και περνάμε στη συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβαστική σε γάμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική D. Δέλτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβαστική ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβαστική F σιγματάφ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβαστική G υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβαστική ας, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβιβαστική η γιώτα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβαστική J, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβιβαστική Κα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβαστική L, ΙΒ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβαστική M, ΙΓ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική N, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβιβαστική Ο, ΙΕ, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Π. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Q. ΙΖ. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Α, Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική R. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική S υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική T υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AV υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική U υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική δι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική X υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Z υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΑ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΒ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΓ AC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΔ ID υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΕ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 32. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική αλφανή. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική αλφαόμικρον. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική AP. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 36. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική AQ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική AR υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική AS υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική AF υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική AG υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G α μικρό υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Ι, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AJ, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AK υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική AL υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική AT υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΜ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στις αναφορές. Μαζί τις ψηφίζουμε την 1 και τη 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο καταπίπτει. 4, 6, 7, 8 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία αριθμός 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 9, 10, 11, 12 μαζί, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα, ερχόμαστε στις νομοδοτήσεις. παράγραφος 22, της Ήτρε, υπέρ, Παράγραφος 10. Απρόκειται για αποκλειστική αρμοδιότητα της ΙΤΡΕ, οπότε δεν ψηφίζουμε εμείς. Δεν έχει αντικείμενο μια τέτοια ψηφοφορία. Ενώ πρέπει να ψηφίσουμε επί της παραγράφου 22. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και έτσι περνάμε στην παράγραφο 2 για την ίντα σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα στην παράγραφο 6 της Επιτροπής Περιφερειακών Υποθέσεων της νομοδότησής της, της ΡΕΓΚΙ, παράγραφος 6. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου με ονομαστική ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. 63 ψήφοι υπέρ, συν μία αν δεν κάνω λάθος για κάποιον που δεν είχε την κάρτα του. Δέκα ψήφοι κατά. Συγχαρητήρια στους δύο συγητές μας. Και έτσι τώρα θα δώσω την προεδρία, παρακαλώ, στον συνάδελφο. Πριν λοιπόν ε, ψηφίσουμε <clears throat> για το κείμενο του κανονισμού, ο κύριος Μπούλμαν έχει στήσει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και εξ ονόματος ε, του συναδέλφου συνεισηγητή του κυρίου Μανουέλου ε. Φερνάντες ε, θα μου επιτρέψετε να κάνω την εξής δήλωση. Και εδώ λοιπόν συνεργαστήκαμε με μεγάλη ομοψυχία. Υπάρχει όμως μία παράγραφος όπου ζητάμε, ετούμεθα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΣΥ, το Steering Board, να ε, αποκτήσει άλλο ένα άτομο, δηλαδή τρεις από την Κομισιόν, ένας που θα εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλος ένας, ένας επιπρόσθετα. Γι' αυτό λοιπόν στο κείμενο αναφέρεται ότι αυτό το επιπλέον άτομο ε, θα ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλες οι πολιτικές ομάδες οι οποίες συμμετείχαν στην επίτευξη αυτού του συμβιβασμού, όλες λοιπόν οι πολιτικές ομάδες δήλωσαν και κατεγράφησαν πρακτικά ότι δεν θα πρόκειται για ευρωβουλευτή, για μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά για μία προσωπικότητα που δεν θα είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που όμως θα προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το λέω αυτό προς αποφυγή κάθε παρεξηγήσεως, ε, μπορείτε να δείτε και τα πρακτικά. Ε, πάντως οι πολιτικές ομάδες μου είπαν ότι είναι καλύπτονται, ότι είναι ευχαριστημένες με αυτή τη δήλωση ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη διευκρίνηση, Λέω ο Πρόεδρος, ε, πάρα πολύ χρήσιμη, το καταγράψαμε στα πρακτικά μας. Και τώρα λοιπόν περνάμε στην ε, ψηφοφορία. Πριν όμως από αυτό πρέπει να πω ότι οι τροπολογίες 295, 153 και 154 αποσύρθηκαν, αλλά θα το επαναλάβω όταν θα φτάσουμε σε αυτές τις ε, τροπολογίες και ξεκινάμε τώρα με την τροπολογία υπερθμών 5-2. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5-3. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική C. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.53 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 2.54 υπέρ, κατά αποχές ε, απορρίπτεται και έμπλ 18 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται έμπλ 19 υπέρ κατά αύριο ε, ψηφίζουμε για την έμπλ 19 παρακαλώ Λοιπόν, συμβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η συμβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η συμβαστική L υπέρ... Α, όχι, αποσύρθηκε, αποσύρθηκε, πάει Είναι αυτή που σας έλεγα προηγουμένως. Η συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβιβαστική, σύβή 321 και M24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική X υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 343. Τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 346 και έμπλη 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 357 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 33 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβαστική N, N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η E, συμβαστική η, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 401 και 402 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 403 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, η H υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται η συμβιβαστική Q. Υπέρ εγκρίνεται η P. Υπέρ εγκρίνεται η κόντ 30 υπέρ απορρίπτεται η 456 υπέρ κατά απορρίπτεται η 457 υπέρ κατά αποχέσει απορρίπτεται, 458 υπέρ κατά αποχέσει απορρίπτεται ή 4... Ρέτζι 39 υπέρ κατά, το ΕΛΚ υπέρ. Η Ρέτζι 39, γι' αυτήν ψηφίζουμε.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 Just a second, we need to check. Okay, so according so so it's covered apparently, so the S&D uh, voting list has a mistake. On... Καλύπτεται. Κάποιο λάθος έχει γίνει εδώ στον κατάλαβο. Η 39 καλύπτεται. Πάμε στην ΙΤΡΕ 45 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η Κόντ 31 υπέρ κατά εγκρίνεται. 468 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική S υπέρ. Σαφές ήταν νομίζω. Θέλετε Μα ήταν σαφές. Η S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 471 και η 472 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 475 υπέρ κατά Τώρα αυτός ο κατάλογος ε, ψηφοφορίας δεν είναι καλός, λέει ο Πρόεδρος. Θα πάρω άλλον. Έχει λάθη ο δικός μου κατάλογος. Συμβαστική D υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, αιτιολογική αναφορά. Η τροπολογία 54, αιτιολογική αναφορά. Η κοντ 1 εγκρίνεται. Η τροπολογία 54 υπέρ. Ο, ακατέπεσε. Η 57 υπέρ κατά απορρίπτεται, η 58 υπέρ κατά απορρίπτεται, η 59 υπέρ κατά απορρίπτεται, η 60 υπέρ κατά απορρίπτεται, η 61 υπέρ κατά απορρίπτεται, η 62 υπέρ κατά απορρίπτεται, η AA υπέρ κατά εγκρίνεται, AB υπέρ κατά εγκρίνεται, AC υπέρ κατά εγκρίνεται, AD υπέρ κατά εγκρίνεται, AE υπέρ κατά αποχές το AF υπέρ εγκρίνεται, AT υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική O, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η συμβιβαστική AG, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η συμβαστική AH, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, AI, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η συμβαστική AJ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η τροπολογία 140 υπέρ κατά εγκρίνεται, η 145 υπέρ κατά απορρίπτεται, η συμβιβαστική AK υπέρ κατά εγκρίνεται, η 154 αποσύρθηκε, πάμε στη συμβαστική AL υπέρ κατά εγκρίνεται, η συμβαστική K υπέρ κατά εγκρίνεται, η συμβαστική AM υπέρ κατά εγκρίνεται, συμβαστική AN υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική A υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική AO υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική AP υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η συμβαστική AQ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η AR συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 214 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική, συγγνώμη, ναι, η συμβαστική AS εγκρίθηκε. Συμβαστική R, υπέρ εγκρίνεται. Η συμβαστική G, υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική U, υπέρ εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ψηφίζουμε τώρα για την πρόταση της Επιτροπής ως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. 65 υπέρ, 11 κατά, 2 αποχές. Και τώρα θα ψηφίσουμε για την απόφαση να ξεκινήσουν διοργανικές ε, διαπραγματεύσεις. Με ονομαστική ψηφοφορία θα ψηφίσουμε παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote is Πέρας 68 υπέρ, 9 κατά, καμία αποχή. Υιοθετείται η έκθεση. Συγχαρητήρια στους εισηγητές και σε όλη την ομάδα. Θα είμαστε πάρα πολύ δυνατοί στον ε, τριμερή διάλογο με τόσο έντονη εντολή. Κλείνει εδώ η συνεδρίαση.